Good afternoon and a happy Καλό σας απόγευμα. Καλή χρόνια σε όλους. Ευχαριστώ που ήρθατε στην συνέντευξη τύπου της Ενωτική Αριστερά. Πρώτα απ' όλα η Γκάμπι Τσίμερ, πρόεδρο τη ομάδα θα λάβει τον λόγο. Μάλιστα. Δεν είναι πια αργά για να ευχηθεί κανεί καλή χρονιά σε όλους και για την καλή συνεργασία. Είναι η πρώτη συνεδρίαση εφέτος στο Στρασβούργο και με την αλλαγή του χρόνου πολλά θέματα σειράξεων ή αντιπαραθέσεων είτε εκ νέου παρουσιάστηκαν ή προσθέθηκαν. Καταρχήν με την Ολλανδική Προεδρία θα ήθελα να ξεκινήσω που αύριο στην Ολομέλεια θα παρουσιάσει το πρόγραμμά της και θα αντιμετωπίσει ακριβώς αυτά τα θέματα και σε αυτά τα θέματα ανήκουν παράλληλα από τα θέματα των τεσσάρων αξώνων που έχουν τεθεί επίκαιρα θέματα που μπορούν να παριθμηθούν όπως για παράδειγμα η εξακολουθούσα σύραξη ή πρόβλημα όσον αφορά τη μετανάστευση το μεταναστευτικό ζήτημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε τον αγώνα, τη μάχη για μια ευρωπαϊκή κοινή λύση που δεν θα συρρυκνώνεται απλά και μόνο να είναι μια λύση στα εξωτερικά σύνορα και ένας μηχανισμός άμυνας κατά πρώτο λόγο και πιστεύω από την άλλη πλευρά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με αυτό το ζήτημα. Και αυτό θα είναι ο πύχης, ο γνώμονας με τον οποίο θα μετρηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά πόσον δηλαδή είναι σε θέση να εκφράσει την αλληλεγγύη της και να ασκήσει τις κοινέ και να εφαρμόσει τις κοινέ αξίες και αρχές της. Ένα δεύτερο θέμα με το οποίο η Ολλανδική Προεδρία θα πρέπει να απασχοληθεί είναι φυσικά η κατάσταση στην Πολωνία που σίγουρα δεν διευκολύνεται με τις αντιπαραθέσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων και της δημοκρατίας ε, της Πολωνίας όπου ο πρόεδρος για παράδειγμα του Συμβουλίου ο κύριος Τούσκ, πρώην πρωθυπουργός της Πολωνίας είναι, έτσι. Και το είδαμε ήδη, το σημειώσαμε ότι μια ολόκληρη σειρά υποδόριων, υποβοσκουσών παρατηρήσεων ε, και ε, θεμάτων αναφύεται. Θέλω ωστόσο για την Πολωνία με ε, ιδιαίτερη προσοχή να αντιμετωπίσουμε τα θέματα θα έχουμε και την ε, Πρωθυπουργό της Πολωνίας. Κανείς στο Ευρωκοινοβούλιο δεν θέλει να χτυπηθεί εντός εισαγωγικών η Πολωνία, να πληγεί η Πολωνία ή να ασκηθούν αυστηρές και οξύες επικρίσεις. Από την άλλη όμως πλευρά παρόλα αυτά η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής <clears throat> για πρώτη φορά όσον αφορά αυτόν τον ε, νέο μηχανισμό που εκπονείται και που τον εξετάζει και τον θέτει υποφώς μια πρώτη κλίμακα εξέτασης θεμάτων που τίποτα άλλο δεν σημαίνει ότι ακριβώς το ζήτημα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν με την Πολωνία σε ένα διαθρωμένο, δομημένο διάλογο. Αυτό ακριβώς χρειάζεται. Διότι προφανώς από αρκετές πλευρές κιόλας με κάποιες μισές αλήθειες ή πληροφορίες ή οξυμένες παρατηρήσεις εργάζονται κάποιοι, αλλά με το πραγματικό πρόβλημα δεν ασχολούνται και το πρόβλημα αυτό δεν την χάνει αντιμετώπιση. Έτσι δεν μπορεί ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε το Συμβούλιο, ούτε κάποιο κράτο μέλο ε, να απεμπολίσει τα θέματα σε σχέση με την Πολωνία και να πει ότι κοιτάξτε μας εξέπληξε αυτή η εξέλιξη, έπεσε εξεθρίας συνέβη. Όχι, δεν συνέβη εξεθρίας. 20 χρόνια είναι, ε, ας το πω έτσι, ε, τα προηγούμενα τα οποία οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση και από το προηγούμενο κόμμα ανταγωνιστικό ε, σύστημα προς την οικονομία, κοινωνική οικονομία της αγοράς υπήρξαν πολλά προβλήματα που αντιμετώπισε ο πολωνικός πληθυσμός ο οποίος αγνοήθηκε ή τέθηκε στο περιθώριο και έτσι λοιπόν δεν πρέπει να εκπλήσεται κανείς γι' αυτό δεν είναι θέμα αρχών ή αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το θέμα του πώς μπορεί να βελτιωθεί η ζωή τους αυτό είναι εκείνο το οποίο τους απασχόλησε αυτό πρέπει να συζητήσουμε είναι χήμερα, είναι αυταπάτη να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να οπισθοδρομήσει η Πολωνία σε ένα νεοφιλελεύθερο καθεστώς με νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση και ότι αυτό θα επέλυε τα προβλήματα της Πολωνίας. Όχι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων που επέλεξε το πίσω, την, το κόμμα αυτό και οδηγηθήκαμε σε αυτήν την εξέλιξη. Δεν μπορούμε να ρίχνουμε στάχτη στα μάτια και να λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ή να το αγνοούμε. Και πρέπει να δούμε τα προβλήματα αυτά και την αντιμετώπιση του συνταγματικού δικαστηρίου και των μέσων του τύπου φυσικά. Και όλα αυτά πρέπει να εξεταστούν. Δεν μπορεί μόνο να συρρυκνώνουμε το θέμα σε, ένα, σε μία αιστεία μόνο. Πρέπει να προχωρήσουμε σφαιρικά. Το τρίτο εξωτερικό πολιτικό ζήτημα που εδώ τουλάχιστον θα τεθεί στο προσκήνιο και υπάρχουν και λόγοι γι' αυτό αναφέρεται στο ότι αύριο θα έχουμε μια συζήτηση στην ημερήσια διάταξη που προβλέπεται από την ημερήσια διάταξη για την κατάσταση στην νοτιοανατολική Τουρκία σε σχέση με τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ερντοάν της Τουρκίας τη συμφωνία που έγινε όσον αφορά το ζήτημα των προσφύγων, η συζήτηση που ε, προχώρησε για την ένταξη της ε, Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών και μετά την αναγνώριση της Τουρκίας ως ασφαλούς χώρας, είπαμε αμέσως ότι αυτό ανοίγει πύλη και πόρτες στον Ερντογάν ο Εντοάν ανεξέλεγκτα, χαλήνοτα, χωρίς επικρίσεις ε, να δράσει κατά των Κούρδων και να πλήξει τους Κούρδους ανεξέλεγκτα. Είδαμε που οδήγησε αυτή η κατάσταση. Είναι μια επίθεση κατά των Κούρδων πολιτών ε, αυτή η στάση του Ερντοάν σε αυτό το τμήμα της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Ζητάμε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και θα το κάνουμε και αύριο να υπομισθούν τις ευθύνες τους, να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους, ε, να μπορέσουν να δράσουν ώστε πρώτον η πίεση στην τουρκική κυβέρνηση να αυξηθεί ώστε άμεσα οι επιθέσεις κατά των Κούρδων, των αμάχων Κούρδων να πάψουν άμεσα οι επιθέσεις αυτές, η ειρηνευτική διαδικασία να, να συνεχιστεί, να ε, ξαναξεκινήσει, οι ειρηνευτικές διαβουλεύσεις για την ειρήνευση και αυτό ανήκει στο ότι αμέσως η κατάσταση ανάγκης η, ε, κατάσταση, η έκτακτη κατάσταση που ισχύει στην νοτιοανατολική Τουρκία πρέπει να σταματήσει η κατάσταση πολιορκίας και πραγματικά ούτε οι υπηρεσίες είναι δυνατόν να διασφαλιστούν ούτε η κάλυψη των αναγκαίων των θεμελιωδών αναγκών των πολιτών ούτε καν η ταφή των νεκρών και όλα αυτά δεν μπορούν να συνεχιστούν και με το σκηνικό του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία Τουρκία θέλει λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση απλά να αποσαφηνίσει τα θέματα των προσφύγων με την Τουρκία και ξεχνά αυτά τα ζητήματα της Νοτιοανατολικής Τουρκίας και των Κούρδων αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και με την Ολλανδική Προεδρία ολοκληρώνοντας δύο σημεία θα ήθελα σύντομα να αναφέρω και να προσθέσω που αναφέρονται στις προτεραιότητες της Ολλανδικής ε, Προεδρίας η Ευρώπη ως ε, αιστεία καινοτομία ε, και απασχόλησης μας εκφλήσει πως θέλει να επιτύχει τον στόχο της η Ολλανδική Προεδρία αναβαθμισμένες θέσεις απασχόλησης να δημιουργηθούν κατά αυτή την περίοδο και ταυτόχρονα να υπάρξουν ριζοσπαστικές αλλαγές ε, της αγοράς ε, και της οικονομίας. Αυτά τα δύο δεν συνάδουν μεταξύ τους, πρέπει να το πούμε. Υπάρχει μια αντίφαση εδώ, εσωτερική αντίφαση που καταδεικνύει ότι από τη μέχρι σήμερα εξέλιξη και από την αυξανόμενη αποχή ή αποστροφή των πολιτών σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται υπεύθυνη για την κοινωνική επιδείνωση δεν έχουν συναρθεί τα αναγκαία συμπεράσματα και μαθήματα από κάποιους. Αυτό πρέπει να το αναφέρουμε σε αυτό το σημείο. Το αναφέρω λοιπόν και για το σημείο για την μελλοντική πολιτική για το κλίμα και την ενεργειακή πολιτική από πλευράς ε, των εκπροσώπων της Προεδρίας αναφέρθηκε ότι 90% ε, της Ολλανδίας βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της επιφάνειας ε, της, της στάθμης της θάλασσας και έτσι ενδιαφέρονται άμεσα αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσουν να προχωρήσουν όπως αναφέρονται και σε ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τα άλλα και τι σημαίνουν όλα αυτά σημαίνουν ότι θα καταβληθούν προσπάθειες η αποδοτικότητα της ενέργειας να αυξηθεί σημαντικά Καθώ καθώς και το τμήμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ανανεώσιμων κατά 30%. Φιλόδοξη στόχη είναι αυτή και θα είναι ένα θέμα αυτό το οποίο αύριο θα το συζητήσουμε και θα το θέσουμε στην Ολλανδική Προεδρία. Αυτά ενημερωτικά από πλευρά μου. Και δίνω τον λόγο σε εσά στη συνέχεια, έτσι. Στον κύριο Χατζηγεωργίου, στον Τάκη, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Η δική μου αναφορά έχει να κάνει με το τι τρέχει στην νοτιοανατολική Τουρκία, όπου εξελίσσεται μια πάρα πολύ τραγική υπόθεση. Έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις τον τελευταίο καιρό ότι είναι πιθανόν η Τουρκία να εξελιχθεί σε μια νέα Συρία με όλα τα τραγικά συνεπακόλουθα και για την Ευρώπη αλλά πρωτίστως βέβαια για τον ίδιο τον λαό της Τουρκίας και τους Κούρδους πολίτες της Τουρκίας. Όταν πριν αρκετά χρόνια ε, είχαμε ονομάσει την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη ως τον παγωμένο αραβικό χειμώνα, μερικοί μας έβλεπαν με θυμηδία, γιατί δεν μπορούσαν να κατανοήσουν την πραγματική κατάσταση στην περιοχή και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε αυτές τις χώρες. Σήμερα, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για τον τουρκικό λαό και ιδιαίτερος της Τουρκίας, εάν δεν ανοίξει τα αυτιά της η Ευρωπαϊκή Ένωση οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συγκρατήσουν <clears throat> αυτό το πρόβλημα, να καταφέρουν να ανοιχθεί ένας ειλικρινής και ουσιώδης διάλογος μεταξύ Κούρδων και τουρκικού κράτους, έτσι ώστε να αποδοθούν στους Κούρδους πολίτες τα δικαιώματα που τους αναλογούν, τότε οι κίνδυνοι να δούμε ένα καινούριο κύμα προσφύγων αυτή τη φορά Κούρδων από την Τουρκία προς την Ευρώπη είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι βεβαίως το μικρότερη σημασία ζήτημα εάν το συγκρίνει κανείς με τις πολλές δολοφονίες ε, απλών πολιτών μέσα στις πόλεις και τα χωριά των Κούρδων στην νοτιοανατολική Τουρκία και βεβαίως με το, μετανάστευση, την μετακίνηση χιλιάδων ανθρώπων από τα σπίτια τους για να αποφύγουν τους ε, κινδύνους που συνεπάγεται η επίθεση του τουρκικού κράτους ενάντια στις πόλεις τους. Ε, συνεπακόλουθο ζήτημα αυτού ε, είναι η ανάγκη ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναδείξει αυτό το ζήτημα στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Είναι μια ευκαιρία η αυριανή συζήτηση η οποία δυστυχώς ε, δεν θα ακολουθείται από ένα ψήφισμα που θα στέλνει τα μηνύματα που θέλουμε το τρίτο που έχω να πω είναι ότι αύριο θα υπάρξει συνεδρία της Μικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στην παρουσία του Τούρκου πρέσβη. Ε, κύριο θέμα θα είναι ε, το κουρδικό ζήτημα και οι επιθέσεις στις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως. Τέταρτο θέμα στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι ότι επήγει μια ε, επίσκεψη ευρωβουλευτών στην περιοχή της των νοτιοανατολικής Τουρκίας έτσι ώστε να καταδειχθεί <clears throat> με τον πιο καθαρό τρόπο το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου. Δυστυχώς όταν έθεσα το ζήτημα αυτό την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες στον κύριο Μπροκ κατά τη διάρκεια συζήτησης της Επιτροπής Εξωτερικών είπε ότι ε, έγινε επίσκεψη την περασμένη άνοιξη ε, και ότι ασκήθηκαν ιδέουσες υποθέτω υποδείξεις ε, προς την Τουρκία για να δοθεί μια λύση στο κουρδικό ζήτημα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν έγινε καμιά επίσκεψη στην περιοχή. Ήταν επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικών στην Τουρκία, αλλά αυτό δεν είχε να κάνει τίποτα με επίσκεψη στην, ε, στις περιοχές στις οποίες αναφέρομαι. Γι' αυτό και προσπαθούμε τώρα να δούμε πώς ε, χωρίς επίσημη αποστολή της Επιτροπής Εξωτερικών να υπάρξει παρόλα αυτά επίσκεψη ευρωβουλευτών από διάφορες πολιτικές ομάδες έτσι ώστε ο αντίκτυπο και το βάρος της επίσκεψης ε, να έχει την, ε, τη σημασία του. Κλείνω με το εξή: <clears throat> Νομίζω ότι η τουρκική κυβέρνηση ε, αισθάνεται ως θανάσιμο τον κίνδυνο της δημιουργίας Συριακού Κουρδιστάν το οποίο θα συνδέεται και γεωγραφικά με το Ιρακινό Κουρδιστάν και αυτό σε συνδυασμό με την αναζωπήρωση ε, της θέλησης των Κούρδων της Τουρκίας για να τους αποδοθούν τα δικαιώματα τους ή και για αυτονόμηση <clears throat> εκλαμβάνει, επαναλαμβάνω αυτή την, αυτό το σύνολο των, των δεδομένων ως κίνδυνο για την ίδια και αντιδρά με έναν τρόπο που υπερβαίνει κάθε έννοια ε, νόμου δικαίου ε, με αποτέλεσμα ε, τις δολοφονίες, ε, τους κατοίκων περιορισμούς ε, των πολιτών της περιοχής αυτής. Γι' αυτό πρέπει να γίνει έκκληση σε ανώτατο επίπεδο προς ε, την Τουρκία να ανοίξει άμεσο διάλογο με τους εκπροσώπους των Κούρδων πολιτών έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί όλα τα βασικά αιτήματα των Κούρδων της Τουρκίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Τάκη ή Κορνέλια Ερνστόρ για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Ναι, να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα από την εξωτερική πολιτική στην εσωτερική πολιτική που όμως είναι εξίσου σημαντική. Ξέρουμε ότι είναι ένα μεγάλο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ψηφιακή ημερήσια διάταξη, το ψηφιακό θεματολόγιο και η ψηφιακή ενιαία εσωτερική αγορά. Μεγάλα βήματα γίνονται, καμιά φορά πιο μεγάλα, καμιά φορά πιο μικρά και μια έκθεση που ε, ψηφίστηκε προς έγκριση που ίσως δεν ήταν τόσο μεγάλης εμβέλειας που αποσαφήνισε όμως κάποια πράγματα για τα οποία θα συζητήσουμε τους επόμενους μήνες και θα αποφασίσουμε 28 ρυθμιστικά πλαίσια υπάρχουν αυτή τη στιγμή από 28 κράτη και ο εναρμονισμός είναι ένας ε, φιλόδοξος στόχος που υποστηρίζουμε. Τα θέματα που εγώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτά και που η ομάδα μας σε αυτά στηρίζεται και προχωρεί και προαγάγει είναι ότι είναι σημαντικό η εσωτερική αγορά αφενός να προχωρήσει αλλά και τα δικαιώματα των πολιτών να είναι σεβαστά. Δηλαδή δεν επαρκεί αν στο ψηφιακό θεματολόγιο για την εσωτερική αγορά ε, εστιαζόμαστε στον ανταγωνισμό μόνο αποκλειστικά. Είναι αναγκαίο και για την ασφάλεια και για την υπολογισμότητα και λογοδοσία να κάνουμε λόγο. Και είναι σημαντικό επίσης όλα τα θέματα τα οποία προτείνονται προς έγκριση να δούμε σε σχέση με την προσωπική ζωή, την ιδιωτική ζωή των πολιτών και τα δεδομένα τους τι θα γίνει με την προστασία τους. Δεν είναι δεδομένα όλα αυτά, δεν είναι εκ προημίου, ε, δεν έχουν αποφασιστεί και ρυθμιστεί και ελπίζουμε ότι θα προαχθούν. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες και αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν θα προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το δεύτερο σημείο που είναι σημαντικό για μας είναι η πρόσβαση και επιχειρηματιών και επιχειρήσεων ισότιμα και ισοδίκαια στην εσωτερική ε, ψηφιακή αγορά. Για την... Δεν πρέπει να υπάρχουν διαφορές και διακρίσεις. Δεν είναι μόνο αναγκαίο αυτό διασυνοριακά, αλλά και από πλευράς προσέγγισης και σύλληψης. Αυτό είναι ένα από τα κέρια θέματα στη συζήτηση για την ψηφιακή εσωτερική αγορά. Σημαντικό είναι επίσης ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι καταναλωτές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχουμε ηλικιωμένους ανθρώπους για παράδειγμα που δεν μπορούν να ενταχθούν ε, ισοπεδωτικά στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των άλλων και πρέπει να δούμε τις ανάγκες αυτές ε, μέσα στο πλαίσιο της ε, ψηφιακής αγοράς. Δεν μπορούν τα πράγματα να παραμείνουν αναλύωτα χωρίς να αλλάξουν. Πρέπει να συνεισφέρουμε να αλλάξει η κατάσταση όσον αφορά τη διαφοροποίηση των αναγκών και για το geo-blocking και τη συζήτηση που ίσως σας είναι γνωστή, η ομάδα μας είπε σαφώς ότι πρέπει να καταργηθεί το geo-blocking <clears throat> διότι είναι άδικες και αθέμητες πρακτικές, οι πρακτικές αυτές του geo-blocking και να σκεφτούμε τι δικαιολογείται και τι όχι σε σχέση με όλες αυτές τις δράσεις από την άλλη πλευρά υπάρχει η πεποίθηση ότι μάλλον παραμένουν ε, οι διακρίσεις εις βάρος μειονοτήτων σε κάποιες χώρες ένα, για παράδειγμα ένας δημόσιος τηλεοπτικός σταθμός δεν μπορεί να δημιουργηθεί λόγω κολλημάτων από, από την άλλη πλευρά λόγω της κύριας μειονοτικής γλώσσας ε, δεν υπάρχει έγκριση και αδειοδότηση και αυτό είναι αρνητική διακριτική μεταχείριση για ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς διότι στερούνται πληροφορίες και εκπαίδευση και παιδεία οι μειονότητες οι άνθρωποι αυτοί. Είναι σημαντικό σε μια εσωτερική αγορά στην, για τους πολίτες μας να διασφαλίζονται τα δικαιώματα στην παιδεία και στην ελευθερία της έκφρασης από πλευράς μέσων του τύπου. Δεν είναι απλά βέβαια όλα αυτά, αλλά πρόκειται για την κατάργηση των διακρίσεων. Το άλλο σημείο είναι ένα άλλο φλέγον ζήτημα η ουδετερότητα του δικτύου. Όλοι λένε ότι χωρίς την ουδετερότητα και αμεροληψία του δικτύου δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Εμείς δεν είμαστε ενθουσιώδεις υπέρ, διότι υπάρχουν προθέσεις και προσφορές για την προσπελασιμότητα στο δίκτυο. Η προσπελασιμότητα πρέπει να είναι χωρίς διακρίσεις συνολικά και για τις προσπάθειες που θα γίνουν για να πετύχουμε κάποια πράγματα στο μέλλον. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες αυτές και υποστηρίζουμε, αποκοινούμε τους πρασίνους αυτή την προσέγγιση. Σημαντικό είναι για μας η διεύρυνση του ευρυζωνικού φάσματος και είναι σημαντικό για τα κράτη-μέλη. Έχει μεγάλη σπουδαιότητα, ιδιαίτερα για τον χώρο της υπαίθρου. Δεν συμμεριζόμαστε την προσέγγιση στην έκθεση ότι κυριότερα πρέπει να εστιαστούμε στους ιδιωτικούς επενδυτές. Όχι, λέμε κοινοτικοί επενδυτές και συνεταιριστικοί συνεταιρισμοί πρέπει να υποστηριχθούν. Μια και στο έργο τους δεν πρόκειται μόνο για το κέρδος, δεν είναι η κερδοφορία η μέρημνά τους, αλλά η κάλυψη των αναγκών των κοινοτήτων. Και εδώ έχουμε και ε, παραδείγματα τα οποία μπορούμε να αναφέρουμε που θα μπορούσαμε με το διευρυζωνικό δίκτυο να υποστηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες αλλά να μην ξεχνάμε επίσης ότι τα κονδύλια από τον ορίζοντα 2020 ως εγχείρημα έχουν περικοπεί. Θα θέλαμε να διασφαλιζόντουσαν αυτά τα κονδύλια και να παρέμεναν αναλύωτα ώστε να χρησιμοποιηθούν για το διευρυζωνικό φάσμα. Και για το Connecting Europe, τη διασύνδεση της Ευρώπης ε, στα, στο διαδίκτυο και στα διάφορα δίκτυα, θα πρέπει να γίνει κάποια προσπάθεια να υπαρκέσουν τα, τα κονδύλια, να καλυφθούν οι ανάγκες και η συζήτηση για την κυβερνοεγκληματικότητα και τα συναφή θέματα είναι θέματα τα οποία ε, είναι ούτως ή άλλως ε, ακαθόδη. Θα πρέπει να μιλήσουμε για εγκληματικότητα σφαιρικά ώστε να καλυφθούν αυτά τα ζητήματα και στη Γερμανία κατά τα άλλα έχουμε και τα θέματα του Google και του Facebook ε, που δημιουργούν προβλήματα και που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να καταργηθούν προνόμια και μονοπόλια και για την ε, διαγραφή σχολείων και παρατηρήσεων μίσους ε, σε αυτά τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και ενημέρωσης ε, πρέπει να γίνουν τα αναγκαία και να καταλήξουμε στο ότι οι εργαζόμενοι που τα δικαιώματα στην εργασία τους πρέπει να προστατεύονται και να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο κουλτούρας και πολιτισμού για αυτά είναι πολύ σημαντικά εγχειρήματα αυτά και προθέσεις και θα πρέπει έτσι να προχωρήσουμε ευχαριστώ Ευχαριστούμε Κονή. Έχουμε πέντε λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις. Μαλή, ε, ε, ε, δημοσιογράφος του Κική Τηλεόραση. Αναφέρατε ότι αύριο δεν πρόκειται να γίνει κάποια γραπτή δήλωση, κάποιο ψήφισμα. Για ποιο λόγο δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Δεύτερον, θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μια ειδική πρωτοβουλία για αυτό το σκοπό και αν ναι, με ποιον τρόπο. Δεδομένου ότι και παλιότερα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε για τη Βόρεια Ιρλανδία είτε για άλλα μέρη του κόσμου. Ευχαριστώ. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με τους ε, πρόεδρους ε, εξετάστηκε αυτό το θέμα για τη συζήτηση να εγγραφεί αυτό το θέμα στην ημερησία διάταξη αυτής της εβδομάδας για την κατάσταση στην νοτιοανατολική Τουρκία και σχετικά γοργά καταδείχθηκε ότι αν θέλουμε να το πετύχουμε αυτό να συζητηθεί δηλαδή αυτό το θέμα αυτή την εβδομάδα αυτό θα ήταν δυνατό μόνο αν δεν επιμέναμε σε ένα ψήφισμα για την αυριανή μέρα. Έχουμε μόνο την ανοιχτή δυνατότητα ως λύση δεδομένου του ότι αύριο θα δοθούν εξηγήσει και δηλώσεις από, το Ευρωπαϊκό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συζητήσει στο Κοινοβούλιο απορρέει από αυτό ότι θα υπήρχε η δυνατότητα ένα ψήφισμα στην επόμενη συνεδρίαση να είχαμε στη συνεδρίαση στην Ολομέλεια μετά από δύο εβδομάδες πάλι εδώ στο Στρασβούργο. Αν θα γίνει αυτό τελεσίδικα και τελικά δεν μπορώ να το προδικάσω. Το πιο σημαντικό για μας ήταν να ανοίξει αυτή η δυνατότητα τώρα που είδαμε ότι μπορεί να ανοίξει. Η κατάσταση στην Τουρκία να συζητηθεί ανοιχτά και δημόσια και το πέπλο της σιωπής να σκιστεί, να διαραγεί. Αυτό ήταν το πρώτο σημείο, η πρώτη προτεραιότητα για να συνεχίσουμε μετά στη συνέχεια να προοδεύσει το θέμα. Ε, η συζήτηση που σε κάποιες χώρες μετά την, το πραξικόπημα, μετά το τρομοκρατικό πλήγμα στην ε, Κωνσταντινούπολη που έγινε δεν πρέπει να αποσιωπηθεί και να οδηγήσει σε σιγή ηχθείως σιγή θανάτου, αλλά θα πρέπει σε σχέση με τον πληθυσμό των κρατών μελών να τους επεξηγηθεί το τι συμβαίνει στην Τουρκία και να υπάρξει πληροφόρηση στον κόσμο για τα θέματα, τα προβλήματα της Τουρκίας. Μπορούμε να μην έχουμε τέτοιες βρώμικες συμφωνίες και ελπίζουμε ότι η κυρία Μέρκελ και οι άλλοι θα συνειδητοποιήσουν τις ευθύνε τους όχι μόνο για τα θέματα των προσφύγων και να ασχολούνται μόνο για την επίλυση κάποιων συμφερόντων τους σε σχέση με τους πρόσφυγες με κύριο σύμμαχο την Τουρκία αλλά δεν μπορεί να υπάρξει αποσιώπηση των επιθέσεων κατά των Κούρδων αμάχων από την τουρκική κυβέρνηση. Αυτό θέλαμε να κάνουμε, να συζητηθούν αυτά ανοιχτά. Ευχαριστούμε Γκάμπη. Υπάρχει άλλη μια ερώτηση από την τσεχική τηλεόραση. Έχω μια ε, ερώτηση για τον Τσέχο Ευρωβουλευτή κ. Άνστορφ που δραστηριοποιήθηκε πολιτικά στην ομάδα σας. Ήθελα να σας ρωτήσω διότι ανακρίνεται για οικονομική απάτη από την Ελβετική Αστυνομία. Θέλω να μάθω αν ακόμη λαμβάνει χρήματα από την ομάδα. Επειδή δεν έχει βγει από την ομάδα, εξακολουθεί να είναι μέλος. Πρακτικά λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιήσει, να, υποφ... έχει όλα τα ωφέλη ως μέλος της πολιτικής ομάδας. Μπορείτε να το εξηγήσετε. Ευχαριστώ. Ναι, με τον Μύροσλαφ Ράμστοφ ο οποίος ε, είχε κατηγορηθεί από ελβετικές αρχές ότι σε μια ελβετική τράπεζα και μάλιστα ε, χαλκευμένα έγγραφα κατέθεσε, πλαστά έγγραφα για να κάνει μια συναλλαγή. Κάτι τέτοιο είναι ασύλληπτο για μένα και ότι ζητήθηκε, λέει, απαιτήθηκε από αυτόν να ακολουθηθεί μια διαδικασία, ζητήθηκε να αποσαφινιστεί από τον ίδιο και να μας πει ποια ήταν τα κίνητρά του και τι κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία και μαζί του λάβαμε την απόφαση ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να αποσαφινιστούν αυτές οι κατηγορίες τις οποίες αρνείται αυτός και απορρίπτει και ως ομάδα αποφασίσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να αποσαφινιστεί κατάσταση. Δεν είμαστε κριτές και δικαστέ. Λαμβάνουμε υπόψη ότι δήλωσε ότι είναι αθώο και θα πρέπει να προστατευτεί η αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας και είπαμε ότι ε, θα πάψει να είναι ενεργό, ενεργά να συμμετέχει στι εργασίες ε, της ομάδα, δεν θα συμμετέχει σε δηλώσεις, ε, δεν θα θέτει αιτήματα για την ομάδα, δεν θα ενεργοποιηθεί για την ομάδα, σταματάει η ενεργοποίησή του και αυτό είναι το θέμα το οποίο υπάρχει εδώ. Τα δικαιώματά του όμως ως βουλευτού δεν περικόπτονται, δεν ε, ε, συρρυκνώνονται. Αν τώρα τα κονδύλια θα καταβάλλονται από εμάς ή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι ο Ευρωβουλευτής έχει δικαίωμα να καταβάλλεται ο μισθός του και να ε, μπορεί να ε, έχει τα χρήματα αυτά στη διάθεσή του. Αυτό όμως είναι πουσιώδες για μένα. Είναι και παραμένει Ευρωβουλευτής. Και αυτό εξαρτάται και συναρτάται και με το τσεχικό δίκαιο και το τσεχικό σύνταγμα. Κάποιος, ακόμα και αν έχει καταδικαστεί δεν ε, χρειάζεται να επιστρέψει να απεμπολίσει την ε, ε, εντολή του. Δεν μπορεί να υποχρεωθεί μέχρι τελικής καταδίκης να επιστρέψει την εντολή του και να αποσυρθεί από την πολιτική ζωή. Και τα θα δούμε τι γίνεται σε σχέση με την ελβετική δημόσια τάξη και το ποινικό δίκαιο. Όχι ότι κάτι καινούριο υπάρχει και παραμένουμε τώρα σε αυτό ότι η κατάσταση αυτή θα αποσαφινιστεί ως έχει. Thank you. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Α, υπάρχει άλλη μια ερώτηση. Παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου ο μιλητής. Sorry. Τόνι Μόμπιν, SC Magazine, Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ ενδιαφέροντα ορισμένα από τα ζητήματα που αφορούν την ε, έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών ασφαλείας και της αστυνομίας. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την επιτήρηση και την ενημέρωση. Θα τους δημιουργεί προβλήματα ε, η πράξη για την προστασία των δεδομένων των πολιτών ε, με την οποία προβλέπεται η προστασία των δεδομένων των πολιτών μα σήμερα. Κόνη. Η Κορνέλια, ναι. Μπορώ να σας πω ότι προχωρά αυτό η δέσμη μέτρων πρέπει να εγκριθεί, να ψηφιστεί προς έγκριση Θεωρούμε ότι είναι ένα σαφές βήμα προς τα εμπρός αυτό, μια πρόοδος, διότι ένας εναρμονισμός στο πλαίσιο τη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων θα διασφαλιστεί προς όφελος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών θα υποφεληθούν όλοι οι πολίτες είναι ένα θέμα, ένα βήμα προόδου Τώρα, το να πούμε ότι είναι η μόνη θετική και ε, ε, εμβέλειας πρόοδος σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία που θα επιτευχθεί τους επόμενους μήνες, δεν ξέρω ακριβώς πότε, όταν μπορέσει να εγκριθεί. Έχουμε τόσες αρνητικές ε, ειδήσει κατά τον τελευταίο καιρό και δεν βλέπω πουθενά κάτι όπου τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να αγωνίζονται προς μια κοινή κατεύθυνση όλοι και όλες να σημειωθεί πρόοδος όπως εδώ για τα ε, θέματα των προσωπικών δεδομένων και το Ηνωμένο Βασίλειο ε, μπορεί να το δεχτεί. Νομίζω υπάρχει, υπάρχει δυνατότητα αυτής της προόδου και είναι θετικό να το δούμε αυτό και να υποχρεωθούν κάποια μέσα, π.χ. Facebook και άλλα, για την, για την επεξεργασία των ε, ευρωπαϊκών θεμάτων να λαμβάνεται υπόψη η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είναι επιτυχία αυτό. Thank you, Ευχαριστούμε, Κορνελία. Νομίζω ότι έχει εξαντληθεί ο χρόνος που είχαμε στη διαθέσή μας. Δράτω με τις ευκαιρίες για να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας και ευχαριστούμε και τους δερμηνείς.